επίτευγμα της ευρωπαϊκής τεχνολογίας και βιομηχανίας και συμμερίζομαι αυτό που είπατε κυρία Γιάλα Σέντερ. Και το λέω αυτό και σαν τέος επίτροπος υπεύθυνο για τη διαστημική πολιτική. Περνάμε στην έκθεση Χάουταλα. Πρόταση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στέφανεκ. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την έκθεση Στέφανεκ. Τέλος. Δεκτή. 569 υπέρ, 72 κατά, 12 απέχουν. Έκθεση Νεγκρέσκου, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή. Έκθεση Αοστρεβίσιους για τη Συμφωνία Σύνδεσης Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνο σας δεν ακούγεστε. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα και αν έγινε σήμερα το πρωί, αλλά δεν ήμασταν πάρα πολλοί βουλευτές παρόντες, θεωρώ ότι είναι κατάλληλη στιγμή να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Βουλής της Μολδαβίας και να ε, ε, του πούμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ ε, για τη χειρονομία αυτή που είχατε και την επίσκεψή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Eh, Εκ νέου καλώς ήλθατε λοιπόν η παρουσία σας εδώ μας προσφέρει μεγάλη ευχαριστήση. Λοιπόν, έκθεση Αουστρελίσιους. Παράγραφος 7. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Άουιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Στο τέλος της παραγράφου θα προσθέσουμε τη φράση που λέει ότι θα στείλουμε μια επιτροπή παρατήρησης στι εκλογές του Νοεμβρίου 2014. Αυτό έχει συμφωνηθεί και με τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Λοιπόν, διαφωνεί κάποιο με αυτή την προφορική τροπολογία, λέει ο κ. Πρόεδρο. Θέτω σε ψηφοφορία πλέον την παράγραφο 7 τροπολογημένη πλέον. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. Παράγραφος 29. Τροπολογία υπαρίθμ 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Στην παράγραφο 31. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική α. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Μετά το L αγγλικό έχουμε την τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το σύνολο της έκθεσης, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Η έκθεση γίνεται δεκτή. Περνάμε τώρα στη σύσταση Αουστρεβίτσιους για τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Δημοκρατία της Μολδαβίας. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Η σύσταση γίνεται δεκτή. Περνάμε τώρα στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Υπάρχει πρόταση ψηφίσματος από έξι πολιτικές ομάδες με μια προφορική τροπολογία στην αιτιολογική α. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι βίες συγκρούσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς συμφωνούμε και να προσθέσουμε ε, ε πάση περιπτώσει, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται πολιτικές ατιμορρησίες. Υποστηρίζουν κάποιοι την τροπολογία αυτή. Υπάρχει και εσύ, φαίνεται ότι είναι πάνω των 40% κατά. Συνεπώ λοιπόν θέτω το αρχικό κείμενο σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το σύνολο του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε τώρα στις ε, τουρκικές ενέργειες που δημιουργούν εντάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. 5. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία. Μετά από την παράγραφο 6 έχουμε την 2 και την 3. Έχουν, η 2 έχει αποσυρθεί. Για την προφορική έχει το λόγο ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας προτείνουμε στο κείμενο της τροπολογίας 3 να απαλληφθεί η απαρίθμηση των χωρών αλλά να διατηρηθεί η αναφορά στο σύνολο της περιοχής. Έχουμε συμφωνήσει με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για την πρόταση αυτή. Ποιοι είναι κατά αυτής της πρότασης. Δεν υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κατά. Θέτω σε ψηφοφορία πλέον. Την τρία τροπολογημένη. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή. στην παράγραφο 10, τροπολογία 1. Τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Αν θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το πρώτο τμήμα της πρώτης τροπολογίας. Ψηφίζετε. La votazione chiusa. Πέρα τη ψηφοφορία. Δεκτό. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της πρώτης τροπολογίας. Άρχεται. La votazione Πέρας. Δεκτό. Στο α κεφαλαίο έχουν την τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Για το Σουδάν τώρα έχω το ψήφισμα των έξι πολιτικών ομάδων, έχω την τροπολογία 1, Ποιοι είναι, ψηφίζουμε ονομα, ε, ηλεκτρονικά για την 1. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. Στην παράγραφο 20 έχω την 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μετά από το F αγγλικό το 3 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στο σύνολό του στο ψήφισμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Le votazioni sono concluse e ora passiamo Τελείωσαν οι ψηφοφορίες. Θα περάσουμε τώρα. Στις επεξηγήσεις ψήφου. Ce ne sono 23.